Η μερίσια διάταξη έχει την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα για τους φορτιστές κινητών τηλεφώνων. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καπάτο, ο οποίος είναι και ο συντάκτης της ερωτήσεως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το θέμα το οποίο συζητούμε είναι προφανέστατο και σαφέστατο. Υπάρχουν περίπου 500 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα που υπάρχουν στην Ευρώπη ενεργά και υπάρχουν 30 διαφορετικοί, 30 διαφορετικοί φορτιστές μπαταριών. Και για ποιου τεχνικού λόγου, κανένα λόγο δεν υπάρχει αυτή τη διαφοροποίηση. Δεν υπάρχει καμία αιτία τεχνική φύσεω. Απλώ είναι μια πηγή κερδοσκοπία ανορθόδοξη από πλευρά των παραγωγών και απ' την άλλη είναι επιζήμιο για το περιβάλλον αυτό, προφανέστατα, διότι λόγω αυτής της παγίδας που εις βάρος των καταναλωτών υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια φορτιστές τηλεφώνων που διασκορπίζονται στο περιβάλλον ε, κάθε δύο-τρία χρόνια υπάρχει κυκλική αναλλαγή αυτών των αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος ο κ. Φερχόγγεν ήδη ε, απάντησε και τάχιστα σε δικό μας ε, ερώτημα που ζητούσε μια παρέμβαση τυποποίησης αυτών των συσκευών και σήμερα είμαστε εδώ για να ζητήσουμε από τον Επίτροπο να μας πει πού βρισκόμαστε, τι εξελίξη είχαμε. Μία διέξοδος ενδεχόμενη είναι της αυτορύθμισης, δηλαδή οι κατασκευαστές των κινητών τηλεφώνων και άρα και των φορτιστών μπαταριών να μπορούν συντομότατα να συμφωνήσουν μεταξύ τους ούτω ώστε να συμφωνούν και να τηρούν μια προδιαγραφή που θα θέσει τέρμα σε αυτή τη γελία και επιζήμια κατάσταση. Να πούμε παρεθείς ότι επίτροπε Φερχόγγεν ότι οποιαδήποτε εγγύηση αυτορύθμισης από πλευράς κατασκευαστών θέλουν να μας δώσουν κατασκευαστέ, ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς, θα πρέπει εμείς να πανεύουμε με, μέσω των νόμων σε περίπτωση που δεν θα αρκεί η απάντηση αυτών των κατασκευαστών. Και αυτή η ρύθμιση δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα κινητά, τους φορτιστές κινητών τηλεφώνων, αλλά και άλλους μηχανισμούς, άλλα μηχανήματα ψηφιακά, για τα οποία υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Έτσι, η Ευρώπη θα μπορούσε, και κλείνω πρόεδρε, θα μπορούσε να επιβάλλει προδιαγραφές που στο τέλος θα μπορούσαν να επιβληθούν και σαν παγκόσμιε διαγραφέ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία όσον αφορά ένα σημαντικό τεχνικό θέμα που είναι σημαντικό για τους ευρωπαίου καταναλωτέ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, χαίρομαι που μπορώ να ενημερώσω τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι όντως ε, υπήρξαν πρόοδοι σε ό,τι αφορά την ε, ε, εναρμόνιση των φορτιστών. Ευχαριστώ τους κυρίους Καπάτο και Μάντες για τη προσπάθεια που έκαναν να συμβάλλουν σε κάτι που επηρεάζει την καθημερινή πραγματικότητα των πολιτών. Συμφωνώ ότι πρέπει να τελειώνει αυτός ο πληθωρισμός των φορτιστών. Τα κινητά πρέπει να έχουν ένα φορτιστή ε, για την επαναλειτουργία τους ε, εκατομμύρια φορτιστές υπάρχουν που επιβαρύνουν άσκοπα το περιβάλλον και δημιουργούν πρόβλημα και στους καταναλωτές. Όποιος αλλάζει κινητό σήμερα πρέπει να αγοράσει και νέο φορτιστή. Ακόμα και διαφορετικά μοντέλα του ίδιου κατασκευαστή συχνά δεν ε, καλύπτονται από τον ίδιο φορτιστή. Το θέμα δεν είναι καινούριο, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η φόρτιση ε, του κινητού δεν είναι απλή διαδικασία. Πριν από λίγα χρόνια η τεχνολογία δεν ήταν έτοιμη να προχωρήσει στην πλήρη διαλειτουργικότητα, εναρμόνιση. Υπήρχαν κυρίως ε, θέματα ασφαλείας, γιατί κατά την φόρτιση του κινητού θα μπορούσε να υπάρξει υπερθέρμανση και έκρηξη. Αυτές οι δυσκολίες εντωμεταξύ ξεπεράστηκαν και πια δεν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι κατά της εναρμόνισης. Έτσι λοιπόν έκανα συγκεκριμένα βήματα για να πείσω τη βιομηχανία να ε, θέσει σε κυκλοφορία ε, ένα φορτιστή, ένα μοντέλο. Ε, είμαι βέβαιος ότι θα κινηθεί γρήγορα ο κλάδος, αλλά εμείς ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα και επουδενή δεν πρέπει να αποκλείουμε και νομοθετική ρύθμιση. Γνωρίζετε ίσως ότι οι χειριστές των δικτύων στο τελευταίο συνέδριό τους στη Βαρκελόνη ανακοίνωσαν ότι θεωρούν ότι από το 2012 τα περισσότερα νέα κινητά που θα χρησιμοποιούνται θα καλύπτονται από έναν ενιαίο φορτιστή. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν αρκεί. Η Κομισιόν θέλει πλήρη εναρμόνιση πάνω στη βάση ενιαίου προτύπου και υποχρεωτικής ε, δέσμευσης της βιομηχανίας ότι θα το κάνει. Η Κομισιόν αναμένει από τη βιομηχανία δεσμευτική συμφωνία με τη μορφή μνημονίου μέχρι το τέλος Απριλίου. Αυτό το μνημόνιο θα πρέπει να υπογραφεί από τους μεγάλους κατασκευαστές των κινητών και θα διασφαλίζει ότι κάθε φορτιστής θα μπορεί να φορτίζει οποιοδήποτε κινητό και οποιοδήποτε κινητό να μπορεί να φορτίζεται από οποιονδήποτε φορτιστή. Η Κομισιόν δεν θα διστάσει να υποβάλει νομοθετική πρόταση αν η ε, βιομηχανία δεν συμφωνήσει ε, εθελοντικά. Θεωρώ ότι και στις ψηφιακές κάμερες ή στα, στις συσκευές MP3 θα λυθεί αυτομάτως το πρόβλημα όταν γίνει το πρώτο ρηξικέλευθο βήμα στα κινητά. Αν δεν συμβεί αυτό και εδώ ε, μπορεί να παρέμβει νομοθετικά και θα χρειαστεί να παρέμβει η Κομισιόν. Η Κομισιόν επίσης ε, ε, στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτω ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τους ε, ομιλητές εκ μέρους των ομάδων, πρώτα απ' όλα από το ΕΛ και τους Ευρωπαίους Δημοκράτες, και Ζούμπη και ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε Φερχόγγεν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα των Κινητών, γιατί από κοινού με το, την Κομισιόν και το Συμβούλιο έχουμε αποφασίσει την δεύτερη συμφωνία για την περιαγωγή, roaming, βρέθηκε καλή απόφαση, θα μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές, είναι καλό αυτό δεδομένη της οικονομικής κρίσης και έχουμε και ε, σε καλό δρόμο το ζήτημα των φορτιστών που νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους πολίτες της Ευρώπης. Ε, οι κλάσεις αποδοτικότητας μπορούν να αναφέρονται στην ετικέτα όπως και στα ψυγεία για να ξέρουμε ε, τις δυνατότητες του φορτιστή. Αυτόματι, ε, αυτόματο κλείσιμο μπορεί να ε, προβλέπεται όταν φορτιστεί δηλαδή το ε, κινητό αυτομάτως να κλείνει ο φορτιστής και είναι επίσης σημαντικό για τα Ινστιτούτα Προτυποποίησης να επεξεργαστούν προτάσεις μετά από προτροπή μας που θα επιτρέψουν τα περαιτέρω. Πιστεύω επίσης ότι καλό είναι να υπάρξει και χρονοδιάγραμμα όπως το ανέφερε ο κύριος Επίτροπος ότι μέχρι τον Απρίλιο δηλαδή να επιτύχουμε μια εθελοντική συμφωνία και μετά να προβλέψουμε την προσαρμογή της τεχνολογίας. Από τη μία πλευρά έχουμε βέβαια τη σύνδεση φορτιστή κινητού. Αυτό με τα τεχνικά πρότυπα μπορεί να ρυθμιστεί και θα δούμε και το κομμάτι της σύνδεσης με την πρίζα, με το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προτάσεων. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πανευρωπαϊκό, αλλά παγκόσμιο και ενδεχομένως και ο ISO, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, μπορεί να ε, βοηθήσει για να βρεθεί παγκόσμια πραγματικά λύση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Η κυρία Τικάου έχει το λόγο για ένα τρίλεπτο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα αφορά πάρα πολλούς καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2009 είναι το έτος της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Αν το πρωτόκολλο συμφωνίας υπογραφεί το πρωτόκολλο εθελοντικής συμφωνίας μεταξύ παραγωγών, κατασκευαστών, κινητών τηλεφώνων, αυτό θα είναι ένα βήμα πρόοδου προς μια εναρμόνιση. Πάνω απ' όλα πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τεχνικές προδιαγραφές κοινέ. Είναι σημαντικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που ασχολούνται και οι φορείς που ασχολούνται με την τυποποίηση να φροντίσουν το ώστε να γίνει μια έρευνα στην αγορά να πετύχουν την τυποποίηση. Θα πρέπει να γίνει και μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση των καταναλωτών διότι δεν αρκεί να υπάρχει μια ετικετοθεσία όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα που θα αναφέρει την, αποδοτη, την ενεργειακή τους αποδοτικότητα θα πρέπει να ενημερωθούν οι πελάτες ή οι καταναλωτές για να μάθουν τι είδη ε, φορτιστών υπάρχουν για τα κινητά τηλέφωνα. Το έτος 2012 δεν είναι μακριά και νομίζω ότι αν οι κατασκευαστές επενδύσουν στο νέο τύπο φορτιστή, τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας εντός των προβλεπωμένων χρονικών ορίων. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και κάτι άλλο. Ήδη στην αγορά υπάρχουν κάποιες συσκευές, κάποιοι φορτιστές, οι οποίοι επιτρέπουν την φόρτιση δύο ή τριών κινητών τηλεφώνων. Ακόμα και αν πρόκειται για κινητά τηλέφωνα διαφορετικής μάρκας. Αρκετά είδη κινητών τηλεφώνων μπορούν να φορτίζονται ταυτόχρονα. Θα πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν περισσότερο στην έρευνα που θα μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα, κυρίως έρευνα που θα αφορά τον τομέα των επικοινωνιών και της πληροφορικής. Έχουμε το, πρόγραμμα, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα που δίνει σημαντικά ποσά για αυτό το σκοπό αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε επενδύσει αρκετά ακόμα σε αυτό το τομέα και, στο πρωτό, και το πρωτόκολλο μεταξύ των κατασκευαστών είναι βήμα προόδου σημαντικό που θα πρέπει να οδηγήσει σε κοινέ προδιαγραφέ. Ευχαριστώ. Η Συμμαχία Φιλελευθέρων για την Ευρώπη, ο κύριος Μάντες έχει το λόγο για ένα τρίλεπτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές και εφόσον θα προτείνουμε κάποια λύση πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι διότι επιτέλους κινούμαστε προ κοινέ ε, προδιαγραφέ για τις φορτιστέ των κινητών τηλεφώνων. Βεβαίω, στα πλαίσια του τη εσωτερική αγορά είναι προφανέ ότι θα πρέπει να αποφύγουμε μια παρέμβαση υπερβολική στην αγορά αλλά θα πρέπει να αφήσουμε τους καταναλωτές να επιλέξουν. Και αν οι καταναλωτές δεν έχουν επιλογή, που και δεν την έχουν τώρα, διότι πρέπει να αγοράζουν ένα φορτιστή πάνω το δικό του τηλέφωνο και δεν πάει με άλλα τηλέφωνα και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Δεν έχουν επιλογή τώρα. Και έδειξε η έρευνα ότι 300 εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται από του Ευρωπαίου καταναλωτέ κάθε χρόνο για να αγοράσουν νέου φορτιστέ ανεξάρτητα από τη τιμή του νέου τηλεφώνου. Αυτό είναι ει βάρο του περιβάλλοντο βεβαίω και το, η ζημιά είναι 300 εκατομμύρια ευρώ και η ενέργεια επίσης σπαταλάται έτσι διότι χρησιμοποιείται πολύ ενέργεια την κατασκευή τηλεφώνων και φορτιστών. Ο κ. Καπάτο και εγώ πριν απευθύνουμε, απευθύναμε επί σειρά ετών αίτηση για να έχουμε κοινέ προδιαγραφέ στον τομέα και γι' αυτό συγχαίρω τον Επίτροπο για τον με τον οποίο προτίθεται να τα ρυθμίσει όλα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω επαφών με τη βιομηχανία που θα πρέπει να καταλήξει κάποια λύση. Εάν δεν βρουν αυτή η λύση, τότε η Ευρώπη θα πρέπει να παρέμβει. Δεν θα πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Θα πρέπει να παρακινήσουμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε να φροντίσουν να βρουν πιο χρήσιμη πρακτική που θα ακολουθήσουν. Και η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή κατά την άποψή μου εδώ και 35 χρόνια δεν υποχρέωσα τη γυναίκα μου να να με παντρευτεί, την έκανα να με διαλέξει. Η επιλογή είναι η καλύτερη λύση. Να παρακινεί κανεί τον κόσμο να αποφασίζει μόνο του. Αυτή τη λύση διαλέξαμε και με τη βιομηχανία. Καλούμε τη βιομηχανία να λάβει τα αναγκαία μέτρα τόσο ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση. Συνεπώς πιστεύω ότι η λύση που διαλέξαμε είναι έξοχη και θα ήταν καλό να εισαγάγουμε μια προδιαγραφή για τους φορτιστές των τηλεφώνων, αλλά πρέπει να κάνουμε το ίδιο και για άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Διότι είναι προφανές ότι όταν μετακινούμαστε, πολύ συχνά βρισκόμαστε με συσκευές που μένουν σε θέση stand-by, καταναλώνουν ενέργεια και έχουμε κάποια ηλεκτρική συσκευή, κάποιο τηλέφωνο, έχουμε ξεχάσει το φορτιστή, μα έχει αποφορτιστεί συσκευή και χρειαζόμαστε να βρούμε κάποιον άλλο, μα βρει κατάλληλο φορτιστή. Είναι μπελά αυτό. Λοιπόν, σωστή προσέγγιση που ακολουθείτε πρέπει να είσαστε πολύ στεναροί έναντι των κατασκευαστών, ε, ούτω ώστε να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση και η λύση στην οποία θα καταλήξουμε ελπίζω να είναι η καλύτερη δυνατή λύση και θα ήθελα να σα συγχαρώ που διαλέξατε αυτή την προσέγγιση. Δεν βλέπω την κυρία Νίμπλερ εδώ. Οπότε θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Και έχω τον κύριο Ρούμπιχ, ο οποίος κάτι θέλει να πει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον Επίτροπο. Υπάρχει το ESB ως τη επαφή που μπορεί να μετασχηματίζει και δεδομένα. Δεν θα ήταν αυτό μια εναλλακτική λύση. Ο Επίτροπος. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, το έχω σημειώσει αυτό κύριε Ρούμπη και ήθελα να το πω μάλιστα. Γι' αυτό είμαι τόσο χαλαρός στο θέμα αυτό και ήρεμος, γιατί δεν πιστεύω ότι δυσκολεύομαι τη ζωή της βιομηχανίας, γιατί το πρότυπο UBS ήδη υφίσταται και όλοι οι εμπειρογνώμονές μου μου λένε ότι το πρότυπο που έχουμε να διαπραγματευτεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα ε, ε, όλες τις συσκευές που μπορεί κανείς να τις έχει στο χέρι και για ε, PCs και για κινητά και οτι, οποιαδήποτε συσκευή χειριζόμαστε με το χέρι και μπορούμε να έχουμε, κρατάμε στο χέρι. Και γι' αυτό, και αυτό είναι και η απάντηση στην κυρία Τικάου, ότι το πρότυπο για το οποίο ρωτάει ήδη υφίσταται στην πραγματικότητα. Επίσης να προσθέσω κυρία Βουλευτή ότι πολύ εντατικέ εργασίες λαμβάνουν χώρα τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα της ενεργειακής κατανάλωσης και η επίπτωση στο περιβάλλον αυτών των φορτιστών. Και θα ασχοληθούμε με όλα αυτά στην πράξη όταν επεξεργαστούμε την οδηγία και την πρακτική της εφαρμογή. Την οδηγία δηλαδή που θα ασχολείται με τα τις συσκευέ που καταναλώνουν ε, ενέργεια και, γιατί, και που θα καλύπτονται από την καινούργια πρόταση. Προς τον κύριο Ρίμπιχ, η αυτόμα, το αυτόματο κλείσιμο νομίζω ότι είναι πολύ καλό και δεν ισχύει μόνο για τη, τους φορτιστές. Είναι ένα θέμα με ευρύτερες προεκτάσεις και ήδη ασχολείται με αυτό η Κομισιόν. Και θα σας ενημερώσω ε, σε εύθετο χρόνο για τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έκλεισε η συζήτηση. Τώρα είμαστε στη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Άρα Λάτφορντ όσον αφορά τι οδηγίες προ τι κοινέ προξενικέ ε, αρχές για τα βιομετρικά στοιχεία όταν εξετάζουν αιτήσει ε, θεώρηση. Για τέσσερα λεπτά το λόγο έχει η η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ πολύ κυρία